Okay, um, Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Από ό,τι φαίνεται συμφωνείτε όλοι, επομένως θεωρείται εγκριθήσα. Ε, δυστυχώς υπάρχουν κάποιες ε, ανακοινώσεις. you Μόλις μου λέει η γραμματεία ότι το σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως, ε, το οποίο θα μας απασχολούσε αύριο, νέα στρατηγική για την πολιτική προστασία των καταναλωτών, έχει μετατεθεί. Um, Εντάξει, με αυτή λοιπόν την τροποποίηση Έχουμε έκτακτη συνεδρίαση για λόγω ακροάσεως με τους, προέδρους της, ε, ε, τους υποψηφίους προέδρους της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής. Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, ε, θα γίνει αυτό την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου το απόγευμα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τους ε, υποψηφίους σχετικά ε, με το Προεδρείο, με το, τη Διοικητική Αρχή μάλλον από τις 2.30 ε, μέχρι τις 3 και 15, 45 λεπτά θα έχουμε μία πρώτη συνεδρίαση και κλεισμένων των θεών και με θυρών και μετά θα έχουμε 90 λεπτά ελεύθερη ανοιχτή συνεδρίαση θα κάνει ε, συστάσεις αύριο το ΕΚΟΦΗΝ στις 4 ε, Οκτωβρίου δηλαδή και ευελπιστούμε ότι ε, θα επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα. Επίσης μου ζητήθηκε να πω δύο λόγια σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο ΕΚΟΦΗΝ 16 και 17 Σεπτεμβρίου καθώς επίσης και την αντιπροσωπεία της, ε, ΕΚΟΦΗΝ, της ε, Επιτροπής μας ΕΚΟΝ ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε τον Σεπτέμβριο. Ε, δεν ε, υπάρχουν ήδη μάλλον κάποιες ε, πληροφορίες στον τύπο. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουν παρούσα στην συνάντηση Εκοφίν και Τίμωθη Γκάιντνερ. Είναι η τρίτη φορά που έχω προσκληθεί να συμμετάσχω σε αυτό το άτυπο, σε την άτυπη συνεδρίαση Εκοφίν. Ε, πρέπει να πω ότι συμφώνησα με την άποψη του Τίμωθη Γκάινερ ότι ε, πραγματικά η κατάσταση στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ ανησυχητική και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να καθησυχαστούν ε, οι αγορές. Και είπα και εγώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες και να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη. Εν τω μεταξύ έχουν γίνει κάποια βήματα προς τα εμπρός όσον αφορά αφορά το, την δέσμη μέτρων ε, για την ε, οικονομική διακυβέρνηση ε, και αργότερα οι αρμόδιοι υπουργοί ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πολιτική συμφωνία στην ΕΚΟΦΗΝ να προχωρήσουν με, την, με τον νομοθετικό συμβιβασμό. Επίσης, σχετικά με την Ευρωζώνη 17 θα πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία φυσικά θα πρέπει να βασίζονται στην καλή βούληση όλων, γιατί η, Ευρώπη δεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελείται από 17, αλλά από 27 μέλη και επομένως υπάρχουν προάγματα τα οποία, ε, και λύσεις που θα πρέπει να γίνουν ε, μέσα από την ενωσιακή πρακτική και όχι σε διακυβερνητικές ε, συμφωνίες. Και οι αξιωματούχοι θα πρέπει να έρχονται και στην Επιτροπή Έκονα έτσι ώστε να ενημερώνουν για τα τεκτενόμενα συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει καλή εφαρμογή της συμφωνίας 21ης Ιουλίου. Αλλά ε, υπάρχει μία αμφιβολία σχετικά με το πόσο γρήγορα και το κατά πόσον θα περάσει αυτή η συμφωνία από όλα τα εθνικά κοινοβούλια και εν πάση περιπτώσει ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας ε, θα πρέπει οπωσδήποτε οι χώρες να βρουν εναλλακτικούς τρόπους έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ η ε, συμφωνία ε, και σύμφωνα με τον Υπουργό Γκάιτνερ θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αντιστάθμισης του μηχανισμού σταθεροποίησης. Επίσης, ε, σχετικά με τα ε, swaps και την, ε, και την διαθεσιμότητα ρευστότητα δολαρίων, είδαμε την κρίση της 15 Σεπτεμβρίου και οπωσδήποτε μας απασχολεί πάρα πολύ. Θα πρέπει οπωσδήποτε στο μέλλον να διασφαλιστεί καλύτερη επικοινωνία με τις διοικητικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό συμφωνήσα, συμφώνησα και εγώ και μάλιστα ανέφερα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επανειλημμένα και σε, πολλές, σε πολλά ψηφίσματα συμφωνήσει με τα ευρωομόλογα, τα Eurobonds. Ε, επίσης ε, έγινε ε, λόγος σχετικά με τις... Crisis Έγινε ε, και αναφορά στις ανοιχτές συναλλαγές, short sellings, ε, καθώς ε, επίσης κατεδείχθη ότι το Κοινοβούλιο θέλει οπωσδήποτε να αποτελεί δομικό μέρος του εποπτικού μηχανισμού. Ε, ε, ο φάκελος ε, του Fast Track Treatment είναι κάτι που μας απασχολεί επίσης. Βεβαίως τεχνικά δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι το κείμενο αυτό υπάρχει, μια και υφίσταται μονάχα στα αγγλικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε συζητήσει κάποια κομμάτια του και είναι γεγονός ότι είναι αρκετά γνωστό το μεγαλύτερο τμήμα του περιεχομένου του και ότι εάν δεν υπάρχει νομική βάση όπως ας πούμε ε, βάση της ε, συνθήκης της Βασιλείας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το Κοινοβούλιο να μπορέσει να προχωρήσει το κείμενο αυτό. Ε, στη συζήτηση που ακολούθησε κατεδείχθη ότι όλες οι, όλα τα θεσμικά όργανα ασχολούνται πάρα πολύ με το θέμα της νομικής βάσης. Όσον αφορά τώρα την ε, αντιπροσωπεία της ε, ΕΚΟΝ στην Ουάσιγκτον, Έχουμε έρθει σε επαφή με τους Προέδρους και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Γερουσία και εκπροσώπους του κλάδου στις ΗΠΑ για να συζητήσουμε με τα θέματα αυτά συζητήσαμε και με εκπροσώπους υψηλού επίπεδου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Τα κύρια θέματα που αντιμετωπίσαμε για η κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών για τη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εφαρμογή τη Βασιλεία 2 και 3, καρύθμιση στον ε, τραπεζικό τομέα, ε, φόροι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ε, αμοιβέ στελεχών, δημόσιο χρέο στι Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαχείριση κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα μετά σε ορισμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια ανάπτυξη, η παγκόσμια διακυβέρνηση για τα χρηματοπιστωτικά, ανισότητε, παγκόσμιε προοπτικέ, μοντέλα ανάπτυξη για την Ευρώπη, και τον Οκτώβριο θα δημοσιεύσει η Παγκόσμια Τράπεζα μία έκθεση για τα θέματα αυτά της παγκόσμιας ανάπτυξης. Επομένως είχαμε εφόλου του επιστητού συζητήσεις και θέλω ευχαριστήσω όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας που ήταν παρόντα εκεί. Αν θέλει κάποιος να ξέρει κάτι περισσότερο, ελάτε σε επαφή μαζί μου και θέστε ερωτήματα. Τρίτο σημείο στην ημέρησια διάταξη είναι η Φορολογική Συμφωνία Γερμανίας-Ελβετίας Α, Ζων Πόλη, θέλεις το λόγο. Α, εντάξει. Όχι σε σχέση με αυτά τα οποία λέχθηκαν προηγουμένως. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είχατε πει ότι εγκρίνεται τη θέση του κυρίου Γκέιτνερ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα προσωπικά να δέχεστε τη θέση του κυρίου Γκέιτνερ, του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι και η άποψη της δικής μου πολιτικής ομάδας στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εμείς κάπου έχουμε βαρεθεί να μας δίνουν μαθήματα άτομα, όπως ο κύριος Γκάιτνερ. Αν το ευρώ έχει μια κρίση η οποία έχει τρομάξει ακόμα και τον κύριο Μπομπάμα, εξακολουθεί να είναι ένα νόμισμα το οποίο έχει υψηλή συναλλαγματική ισοτιμία. Οι αγορές δεν μπορούν να υπερτιμούν και να αναβαθμίσουν ένα νόμισμα το οποίο είναι σε τόσο κακή θέση όπως λέει ο κ. Γκάιτνερ. Εγώ δεν υποστηρίζω λοιπόν τη θεωρία συνωμοσία, αλλά από την Αμερικάνικη πλευρά κάνουν ό,τι μπορούν οι Αμερικάνικες ε, τράπεζες ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες να αγοράσουν ευρώ και θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα γύρω από το ευρώ. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα στην Ευρώπη, αλλά τα χρέη αυτά δεν έχουν δημιουργηθεί σε δύο μέρες. Υπάρχουν σημαντικά χρέη κρατικού χαρακτήρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, τουλάχιστον ένα τμήμα της Επιτροπής, το οποίο εκπροσωπώ εγώ, είναι ότι η κατάσταση είναι μεν σοβαρή, αλλά δεν είναι μια κατάσταση για την οποία εμείς θα πρέπει να ζητάμε συγγνώμη από τις ΗΠΑ και από τον κύριο Γκάιτνερ. Uh, Ευχαριστώ, Jean Paul. Εγώ δεν συμφώνησα φυσικά με όλα αυτά τα οποία είπε ο κ. Γκάιτνερ, ο Τίμωθη Γκάιτνερ, αλλά συμφώνησα στο ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέψουμε καταστροφικές ε, εξέλιξεις. Και σκέφτηκα ότι η ιδέα της απομόχλευσης και του να φύγουν τα τοξικά ομόλογα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα, θεωρούσε ότι αυτό είναι μια <clears throat> θετική ιδέα. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ε, Φορολογική Συμφωνία Γερμανίας-Ελβετίας. Εδώ υπάρχει ένα προφορικό ερώτημα, το οποίο έτυχε συμφωνίες μεταξύ μας. Ανταλλάξαμε email σε σχέση με το ποιο θα πρέπει να προσυπογράψει αυτή την προφορική ερώτηση. Εφόσον είναι εξ τη της Επιτροπής μας, εγώ προτείνω να υπογράψω εγώ εξ τη της Επιτροπής μας. Αν θέλουν να υπογράψουν εκεί οι συντονιστέ, τότε θα πρέπει να το κάνουν εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Νομίζω ότι η σωστή αντιμετώπιση προς το παρόν είναι να υπογράψουμε την προφορική ερώτηση ως Επιτροπή, γιατί αυτή είναι η βάση επί της οποίας συμφωνήσαμε για αυτή την προφορική ερώτηση. Αυτό νομίζω ότι είναι πιο φυσιολογική μέθος. Αρλίν, προφανώς. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τη συμφωνία Γερμανίας-Ελβετίας, αλλά αναφέρεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συμφωνία που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ελβετία. Δεν ξέρω γιατί ο τίτλος λοιπόν αφορά μονάχα τη Γερμανία. Ίσως θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη διατύπωση. Και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάνει μια συμφωνία. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρονται και οι δύο χώρες αυτές ή τουλάχιστον να είναι δύο χωριστές προφορικές ερωτήσεις, αν θέλετε. Βολφ Κλίντς. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι σχετικά με την Ελλάδα. Σύμφωνα με ορισμένε πηγές, περίπου 500 με 600 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα είναι καταθέσεις ιδιωτών Ελλήνων. Και το πιθανότερο είναι ότι δεν έχουν φορολογηθεί. Οπότε η Ελλάδα χάνει έσοδα. Θα ενθάρρυνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά να το εντάξει και αυτό στο λεγόμενο πρόγραμμα διάσωσης να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις και η Ελλάδα με την Ελβετία για να μπορέσει να πάρει αυτά που της οφείλουν ως φόρο οι καταθέτες εξωτερικού. Κοιτάξτε, ε, δεν θέλαμε να γίνει συζήτηση. Ζητήσαμε τις προτάσεις σας. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να τα προσθέσω και να αλλάξω τον τίτλο, αλλά θα πρέπει να κατατεθεί σήμερα, εάν πρέπει. Σφεν, Γκίγκολτ. Ένα σχόλιο μόνο. Η διαφορά είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι το κείμενο της Γερμανικής Συμφωνίας είναι γνωστό, ενώ η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί. Οπότε είναι και πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Είναι τεχνικό βέβαια το σχόλιο που κάνω, αλλά ε, επί της ουσίας βεβαίως θα μπορούσαμε να διευρύνουμε το πεδίο. Αλλά όπως σας είπα, τεχνικά η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ακόμα γνωστή. Η ε, Πρόεδρος. Ναι, ξέρουμε ότι κάτι τρέχει όμως. Θα μπορούσαμε να πούμε γερμανική, γερμανοελβετική, ε, φορολογική συμφωνία και άλλες συμφωνίες. Σας είπα ότι δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα της ημερησίας διάταξης και θέλω να προχωρήσουμε. Μπούλμαν, θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό που προτείνει η Αλήν Μακάρθη. Κάτι λέει κυρία Μακάρθη εκτός μικροφώνου. Ähm, Λέγα λοιπόν ότι υποστηρίζω τη διεύρυνση του κειμένου γιατί ο Σφέν Κίργκολτ είχε την καλοσύνη να το πει στην προηγούμενη συνεδρίαση των συντονιστών, να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε τι γίνεται. Με παράδειγμα τη Γερμανική Συμφωνία, την Αγγλική Συμφωνία, τι γίνεται με τις διμερείς συμφωνίες να μην υπονομεύουν την ευρωπαϊκή συνεργασία. Και ε, κάποια στοιχεία που ανέφερε και ο Βόλφ θα μπορούσαν να μπουν ε, ε, στο κείμενο, όπως και η διεύρυνση του τίτλου που είπε η Το υποστηρίζουμε και κατά τα άλλα δεν έχω κανένα πρόβλημα να προχωρήσουμε όπως προτείνετε εσείς. Right. Well, we'll circulate a final draft, seeing if we can sweep up these. Θα κυκλοφορήσει ένα τελικό σχέδιο για να δούμε αν μπορούμε να εντάξουμε και αυτά τα θέματα. Αν χάσουμε όμως την προθεσμία, χαιρετίσματα. Θα μισολαβήσει και άλλη ολομέλεια και δεν θα μπορέσει να εγγραφεί στην της διάταξη. Λοιπόν, θέλω να περάσω στο σημείο 4 τώρα, αναλλαγή απόψεων με το Hans Hocherwurst, πρόεδρο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Γνωρίζω ότι έχουμε καθυστέρηση 25 λεπτών, μας είπε ότι δεν μπορεί να παραμείνει. Αλλά θα ε, αφήσω ε, λίγο χρόνο παραπάνω αν δεν καλύψουμε το χρόνο μας. Ζητώ συγγνώμη. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, thank you Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να σας πω και εξ ονόματος του Φιλίπ Νταζού, του Γάλλου συναδέλφου, ότι είναι χαρά μας βεβαίως το γεγονός ότι βρισκόμαστε ενώπιό σας και ευκαιρία που έχουμε να μιλήσουμε στην ε, τόσο σημαντική σας επιτροπή Μερικοί από εσά ίσω να γνωρίζουν ότι είχα μακρά πολιτική καριέρα στι κάτω χώρε μέχρι πριν από πέντε χρόνια που εγκατέλειψα την πολιτική και χαίρομαι που ξαναβλέπω κοινοβούλιο. Και η υπέρβαση του χρόνου είναι κάτι που θυμάμαι πάρα πολύ καλά και από το κοινοβουλευτικό μου παρελθόν, οπότε δεν με εκπλήσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ενώπιόν σα και με χαρά απαντήσω τι όποιε ερωτήσει που σίγουρα θα έχετε. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιε αγωγικέ παρατηρήσει για δύο βασικά θέματα. Καταρχά, θα ήθελα να πω ε, δύο λόγια για τη σημασία ε, των σχέσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με την Ευρώπη και κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα να σας δώσω μερικά σχόλια και παρατηρήσεις ε, ως προς τα λογιστικά πρότυπα και τη χρηματοπιστωτική κρίση την οποία βρισκόμαστε ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτον, σχέσεις λοιπόν του Συμβουλίου μας με την Ευρώπη. Είναι στρατηγικής σημασίας και για τους δύο φορείς πιστεύω. Η Ευρώπη έχει επενδύσει πολύ κεφαλό και πολιτικό και οικονομικό στην απόφαση της ε, να εγκρίνει το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αγοράς το 2005. Ε, το Συμβούλιο μας ε, με αυτόν τον τρόπο είναι στο δρόμο για να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στη χάραξη προτύπων. Εσείς το εγκρίνατε με μεγάλη πλειοψηφία 458 ψήφων. Επίσης το ε, Κοινοβούλιο ζήτησε το διεθνές πρότυπο να είναι η παγκόσμια κοινώς αποδεκτή γλώσσα ε, για τη λογιστική παγκοσμίω. Αυτή η δράση, για, η κλίση μάλλον για παγκόσμια δράση, ε, της ακούστηκε όλο και περισσότερες χώρες ακολούθησαν να, ε, την Ευρώπη και μέκριναν τα πρότυπα αυτά. Στην Αμερική, Βόρεια και Νότια, σχεδόν Ολόκληρη Λατινική Αμερική και ο Καναδάς συμμετέχει. Στην Ασία, Οκεανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κορέα, Χονγκ και Σιγκαπούρη και προσεχώς η Ινδονησία ε, θα υιοθετήσουν πλήρως αυτό το σύστημα. Η Ιαπωνία επιτρέπει σε κάποιες εταιρείες της να ακολουθήσουν ήδη αυτά τα πρότυπα, ενώ η Κίνα είναι καθοδόν και πολύ κοντά ε, στο να ακολουθήσουν το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αγοράς. Επίση και η Νότια Αφρική και το Ισραήλ συμμετέχουν πλήρω Στην Ευρώπη, εκτό ευρωπαϊκή Ένωση. η Τουρκία υιοθέτησε πλήρω τα πρότυπα και η ε, Ρωσία είναι καθοδόν. Από φέτος η πλειοψηφία, η πλειονότητα των ε, κρατών ε, του G20 χρησιμοποιούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και μάλιστα οι G20 υποστηρίζουν πλήρως τη σύγκληση των λογιστικών προτύπων για να φτάσουμε σε ένα κοινό παγκόσμιο πρότυπο τύπο. Όπως γνωρίζετε, η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς ε, θα αποφασίσει ε, προσεχώς αν θα ενσωματώσει το διεθνές πρότυπο στα δικά της λογιστικά συστήματα και αν το κάνει αυτό με ποιο τρόπο θα γίνει. Θα είναι δύσκολη αυτή η απόφαση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είμαι αισιόδοξο ότι θα ευδοκιμήσει ε, μια αρνητική απόφαση, την οποία ειλικρινά δεν περιμένω, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση μετά από τόσα χρόνια ε, που αφιερώσαμε για τη σύγκληση παγκοσμίω. Μια τέτοια απόφαση, θα σας έλεγα, όσο πίθανη κι αν είναι, θα καθυστερήσει την πρόοδο που έχουμε επιτελέσει, διότι πολλές χώρες αναμένουν να δουν τι θα κάνουν οι ΗΠΑ. Η Ιαπωνία, η Ινδία, και η Κίνα, ε, επί παραδείγματι. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να οδηγήσει σε μεγάλη καθυστέρηση της εργασίας μας. Πιστεύω όμως ότι τώρα έχει αποκτήσει μια δυναμική αυτή η προσπάθεια τόσο ισχυρή που δεν ε, μπορεί ε, πλέον να σταματήσει. Μπορεί να καθυστερήσει, αλλά όχι να σταματήσει. Είναι πάρα πολύ ισχυρή και πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια και δεν έχει επιστροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διαδραματίσει εδώ πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι λοιπόν αξιοσημείωτη η πρόοδο που έχει τελεστεί τα τελευταία δέκα χρόνια η στρατηγική τη Ένωση να δείξει διεθνή ηγετική στάση δικαιώθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το δικό μας Συμβούλιο θεωρεί την ευρωπαϊκή υποστήριξη δεδομένη. Γι' αυτό το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έρχεται σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους ε, όταν εκπονεί τα νέα λογιστικά πρότυπα. Είμαστε σε συνεννόηση και πολύ στενή με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΦΡΑΚ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης και ε, με όλους τους ε, ενεχομένους, τους επενδυτές και άλλους φορείς του κλάδου. Παρά ε, την ένταση και τη συχνότητα των επαφών και του διαλόγου, βεβαίως μπορεί να υπάρξουν μερικές φορές που διαφωνούμε. Η Ευρώπη ενδιαφέρεται κυρίως για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ το Συμβούλιο μας θα πρέπει να ε, ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα όλων ε, παγκοσμίω. Πολλές φορές ε, υπάρχουν και διενέξεις ή διαφωνίες για τα λογιστικά ε, μεταξύ ε, των ίδιων των ευρωπαϊκών κρατών ή μεταξύ επενδυτών και λογιστών. Θα πρέπει εμείς στο Συμβούλιο μας λοιπόν να αποδείξουμε ότι οι επιλογές μας βασίζονται σε καλή απόφαση, καλώς ενημερωμένη, με σωστή γνώση των διαδικασιών και εποπτεία του κλάδου. Επίσης θέλουμε να τονώσουμε την εμπιστοσύνη εκείνων που έχουν υιοθετήσει τα πρότυπά μας. Θα ενισχύσουμε τις θεσμικέ μας σχέσεις με την Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Εμείς μια ανεξάρτητη αρχή που ορίζουμε ε, πρότυπα θα πρέπει να ε, βασιζόμαστε στην εμπιστοσύνη σας. Μπορεί να είμαστε ανεξάρτητοι αλλά δεν είμαστε και ελεύθεροι σκοπευτές. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις είναι το θέμα της χρηματοπιστικής κρίσης και των προτύπων λογιστικής. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι φυσικά έχω στη διάθεσή μου σε αυτές τις στιγμές. Πιστεύω όμως ότι ένα γενικότερο πλαίσιο θα μπορούσε να μας βοηθήσει για να έχουμε μια καλή συζήτηση για το θέμα αυτό. Αυτό που προκάλεσε την κρίση ήταν και η κατάρρευση των επιχειρηματικών προτύπων και η αποτυχία των μακροοικονομικών πολιτικών σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια, αστοχίες της ρύθμισης οδήγησαν τις μεγάλους κινδύνους να διονγκωθούν χωρίς να υπάρξει κάποια αντιμετώπιση τους μέχρι ότου ήταν πολύ αργά. Σε πολλές περιπτώσεις ήταν ανεπαρκής η διαφάνεια για να μπορούν να ξέρουν οι επενδυτές ποιοι ήταν οι κίνδυνοι τους οποίους αναλάμβαναν. Και τη στιγμή που είμαστε στη μέση της κρίσης μπορούμε να πούμε ότι είναι απίστευτο ότι έγινε κάτι τέτοιο και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξαναγίνει. Και από αυτή την άποψη οι χρηματοπιστωτικές εκθέσει έχουν να κάνουν ένα σημαντικό, παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Η διαφάνεια είναι αυτό που ξυπνάει τον αγωγιάτη, δηλαδή τον λογιστή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πολύ σημαντική για μα. Ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνεια θα επιτρέψει αυτού οι οποίοι διαβάζουν του οικονομικού λογαριασμού να καταλαβαίνουν και τι πιο σκοτεινές πτυχέ της οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Η διαφάνεια είναι η μεγαλύτερη συμβολή που μπορούν να κάνουν οι λογιστές στη μακροχρόνια σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η διαφάνεια είναι προαπαιτούμενο για τη μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Χωρίς τη διαφάνεια, τα μέσα τα οποία στοχεύουν σε αυτή τη σταθερότητα είναι απλώς μια φενάκι και επιτρέπουν τη διόγκωση των κινδύνων μέχρι ότου είναι πολύ αργά. Και συμφωνώ βέβαια ότι η διαφάνεια δεν ωρεοποιεί πάντα τα πράγματα. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε επίπεδο διακυμάνσεων και αστάθειας έχουν βαθιές ρίζες. Ο πρόεδρος της Deutsche Bank, ο κύριος Άκερμαν, είπε πρόσφατα ότι η αστάθεια είναι η νέα φυσιολογική κατάσταση. Και πιστεύω ότι οι εποχής που μπορούσε κανείς να κρατάει στοιχεία ενεργητικού χωρίς κανένα κίνδυνο που οι επενδυτές θεωρούσαν ότι κάποιες επενδύσεις είναι απόλυτα ασφαλείς έχουν περάσει αυτές τις μέρες για πάντα. Αν λοιπόν η αστάθεια είναι η νέα πραγματικότητα, πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό από αυτούς οι οποίοι θέτουν τα πρότυπα για τη λογιστική απεικόνηση θα πρέπει να εμποδίσουμε τεχνητά τους επενδυτές να γνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα της αστάθειας ή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε ως το δυνατόν σαφέστερα και με πλήρη διαφάνεια αυτή τη νέα πραγματικότητα. Οι περισσότεροι με τους οποίους μιλώ λένε ότι οι οικονομικές εκθέσεις θα πρέπει να απεικονίζουν την πραγματικότητα όπως είναι. αυτό είναι και ο σκοπός τους εξάλλου. Και όχι όπως θα έπρεπε να θέλαμε να είναι τα πράγματα αν είναι τσίτσιδρος ο αυτοκράτορας, τότε αυτό είναι και η ευθύνη των οικονομικών ελεγκτών να το πούν αυτό, όσο και δυσάρεστο να είναι αυτό, ως αλήθεια. Υπάρχει όμως και μια, ένα σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε εδώ και να το έχουμε υπόψη μας. Όταν ζητάει κανείς από τους λογιστές να παρουσιάσουν την αλήθεια, αυτό είναι, είναι μια άποψη, αλλά συγχρόνως δεν θα πρέπει η ίδια η πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων να προκαλεί περαιτέρω αυστάθεια. Γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο μας έχει κρατήσει πάντα μια πραγματιστική στάση σε σχέση με το ποιε μεθόδους μέτρησης θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μία μονάχα σωστή απάντηση. Και γι' αυτό πάντα ακολουθήσαμε μια προσέγγιση με μικτές μεθόδους, η οποία ε, συνδυάζει την ιστορική λογιστική, δηλαδή βάση του ιστορικού κόστους, με την τιμή αγοράς. Και γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε κάνει μια μεταρρύθμιση των στάνταρ μας για την καταμέτρηση της λεγόμενης fair value της τιμής αγοράς για να έχουμε και μια νέα κατεύθυνση για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που είναι σε αγορές οι οποίες δεν έχουν ρευστότητα γιατί είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις αγορές να καταμετρήσει κανείς την τιμή αγοράς. Γι' αυτό προχωρούμε με επιφυλακτικότητα στη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών εργαλείων και της λογιστική. Οι κανόνες μα για, ε, για τους λογαριασμούς αντισταθμίσματος, hedge accounting, θα έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν αστάθεια για τις εταιρείε οι οποίες θέλουν να αντισταθμίσουν του κινδύνου τους. Δεν πρέπει εμεί να αποκρύπτουμε την αστάθεια, όχι να το πω αλλιώ. η λογιστική δεν πρέπει να αποκρύπτει την αστάθεια, αλλά δεν πρέπει να είναι και η πηγή της αστάθειας. Εν κατακλείδη μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαίρομαι για την προσοχή σας. Είναι φανερό ότι ζούμε σε πολύ ενδιαφέροντες καιρούς. Υπερβολικά ίσως από ό,τι νομίζω και εγώ. Πρέπει όλοι να εργαστούμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε τα βαθιά προβλήματα τα οποία μαστίζουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εγώ είμαι απόλυτα δεσμευμένος μαζί σας ότι η ομάδα μας θα συνεχίσει, το φορές μα, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκομένους και μεταξύ αυτών την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Θέλουμε να βρούμε ευκαιρίες για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μαζί σας και να βοηθήσουμε να αυξηθεί και πάλι η εμπιστοσύνη των επενδυτών στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Πολλά θέματα δεν πρόλαβα να τα αντιμετωπίσω σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση, αλλά είμαι στη διάθεσή σα για οποιαδήποτε ερωτήματα θέλετε να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Thank λέει Πρόεδρος. Would members who Τα μέλη τα οποία θέλουν να θέσουν ερωτήματα θα μπορούσαν να το αναφέρουν. Ο Βόλφ. Βόλφ, πρώτος εσύ. Κύριε Χόχενφορς θέλω να σας ευχαριστήσω φυσικά για την παρουσία σας. Γνωρίζετε πολύ καλά, φαντάζομαι, ότι οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον φορέα σας δεν ήταν πάντα αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς να έχουμε. Πάντα θέλαμε να υπάρχει ένας διάλογος σε τακτά διαστήματα. Αλλά βλέπουμε ότι ο φορέας σας, το, Συμβούλιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ακολουθεί περισσότερο τα αμερικανικά τεκτενόμενα και όχι τα ευρωπαϊκά. Και δεν έχουμε, όπως είπα, αυτό το τακτικό διάλογο που θα είχαμε επιζητήσει. Ελπίζω ότι έχετε δίκιο κατά τα άλλα όταν λέτε ότι είσαστε σίγουρος ότι οι Αμερικανοί θα μπορέσουν να εγκαθιδρύσουν αυτά τα νέα πρότυπα. Έχουμε ακούσει τέτοιες αισιόδοξε δηλώσεις στο παρελθόν και έχουμε απογοητευτεί στη συνέχεια. Ελπίζω λοιπόν θα γίνει πραγματικότητα αυτό. Έχω τώρα ένα καθαρά τεχνικό ερώτημα να σας θέσω. Και επειδή είναι τεχνικό ερώτημα μπορείτε εσείς να το απαντήσετε με συγκεκριμένο τρόπο το ISB, το Συμβούλιο για τα Λογιστικά Πρότυπα, παρουσίασε ένα σχέδιο τον προηγούμενο ε, Ιούνιο σε σχέση με την καταγραφή των εσόδων από συμβόλαια με πελάτες. Και βάσει αυτής της συμφωνίας θα έπρεπε να καθιδρυθεί μια συμφωνία για την απόκτηση εσόδων με, κατά περίπτωση και από θηγατρικές εταιρείες λοιπά. Και σε, στη δική μου περίπτωση στη Γερμανία και ο Ζαν Πιέρ Ζες και άλλοι συνάδελφοι στην Ισπανία έχουν δει τις απόψεις εταιριών, όπως είναι οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών, που λένε ότι αυτό το σχέδιο ουσιαστικά επιτυγχάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτά τα οποία είχαν ζητήσει αυτοί οι ίδιοι. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι δυνατόν να καταγραφούν μελλοντικά έσοδα, έσοδα δηλαδή από μελλοντικά χρόνια βάσει αυτής της ε, αντιμετώπισης των λογιστικών εσόδων. Και αν αυτό έχει να κάνει με το θέμα που ότι οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών πολλές φορές κλείνουν συμβόλαια τα οποία δίνουν επιδοτούμενα τιμολόγια στους καταναλωτές και θέλουν αυτές τις τιμές, το τμήμα λοιπόν που είναι η επιδότηση, να το καταγράψουν αμέσως στα έσοδά τους και όχι να το καταγράφουν στα επερχόμενα έτη. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώς το έχετε δει το θέμα αυτό και πώς θεωρείτε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλίντσα για την ερώτησή σας. Ξέρετε ότι και ε, ο ίδιος ο πρόεδρος δεν είναι ε, αγγλοσαξονικής καταγωγής. Έχω κάποιους αγγλοσάξονες, αλλά δεν είναι και τόσο κακοί, ξέρετε. Είμαστε πολλά, τα... Είμαστε πολλά άτομα, ε, προερχόμαστε από διαφορετικές κουλτούρες και από ε, διαφορετικούς ε, πολιτισμούς, από τις τέσσερις γωνίες του κόσμου. Έχουμε ανθρώπους από την Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καθένας μπορεί να βλέπει, να έχει διαφορετική οπτική γωνία, αλλά παρόλα αυτά όλοι μας και το προσωπικό μας έχουμε ένα μονάχα μέλημα, να προστατέψουμε τα συμφέροντα των επενδυτών ε, και ε, δεν μιλάμε μονάχα για μεμονωμένα άτομα που προσπαθούν να αυξήσουν την προσωπική τους περιουσία. Ε, το θέμα των ΗΠΑ και το κατά πόσον θα εγκρίνουν αυτά τα πρώτα τύπα. Ε, δεν ωφελεί να είμαι απεσιόδοξος, θέλω και οφείλω να είμαι αισιόδοξο. Νομίζω ότι εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε συμφωνήσουν, προσυπογράψουν τα πρότυπα αυτά, θα είναι καλό για όλους και θα πείσουν και κάποιε πιο σκεπτικέ αγορέ, αγορέ οι οποίε είναι ακόμα πιο διστακτικέ. Θα κάνει καλό σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρο το εμπόριο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν πάντοτε πολύ ε, σημαντικό βασικό στοιχείο στην, στα διεθνή λογιστικά και στον καθορισμό διεθνών λογιστικών ε, προτύπων. Ε, όπως είπα και προηγουμένως, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή και με την ε, Επιτροπή, Χρηματοοικονομικής, Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς των πολιτειών. Λοιπόν, εγώ έγινα πρόεδρος πρόσφατα, όπως ξέρετε, και ένα από τα πρώτα, τις πρώτες συναντήσεις ε, που έκανα ήταν, αφορούσε ακριβώς αυτό το θέμα των τηλεπικοινωνιών. Πολλοί πελάτες όταν υπογράφουν ε, συμφωνία με τις ε, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών παίρνουν ένα τηλέφωνο δωρεάν, μια συσκευή δωρεάν και νομίζω ότι ούτε ένας δεν πιστεύει ότι πραγματικά είναι δωρεάν αυτή η συσκευή γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή σε ένα σε δύο χρόνια θα χρειαστεί να πληρώσουν την συσκευή ε, αυτή. Και επομένως μιλάμε για πώληση και είναι πώληση η οποία θα πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν είναι δυνατόν να θεωρήσει κανείς ότι αυτή η συσκευή είναι απολύτως δωρεάν και ότι δεν αποτελεί ε, συναλλαγή εμπορική. και νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να έχει άγνοια της οικονομικής πραγματικότητας για να πει ότι πραγματικά αυτή η τηλεφωνική συσκευή είναι ε, ε, δωρεάν. Ε, βεβαίως αυτές οι εταιρείε ε, θα ε, θέλουν να ξανασυζητηθεί το θέμα. Θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε, να το ξανασκεφτούμε. Και εάν τα επιχειρήματά τους είναι τρομερά και μας πείσουν ότι πραγματικά αυτές οι συσκευές βάσει συγκεκριμένων τιμολογίων είναι δωρεάν, τότε θα αλλάξουμε και εμείς τη θέση μας. Ζωάν Πολ για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για να ολοκληρώσω την ερώτηση του συναδέλφου ε, που ήταν πραγματικά πολύ σκόπιμη, θα ήθελα να επανέλθω στο ίδιο θέμα. Καλό είναι να γίνονται πρότυπα, αλλά θα πρέπει να είναι και οικονομικά ωφέλιμες. Θυμούμε το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ε, για, την, ε, για τον κανονισμό 17 ε, σχετικά με τις EIS 17 σχετικά με την ενοικίαση και έπρεπε να γίνει λογιστικός υπολογισμός για όλη την περίοδο κατά την οποία ας πούμε ενοικιάζουν τα τα γραφεία τους ε, ε, μια εταιρεία, αλλά αλλά όταν αξιολογούν την εταιρεία οι οργανισμοί αξιολόγησης τελικά δεν λαμβάνουν υπόψη τους ε, με τον ίδιο τρόπο αυτόν τον υπολογισμό. Η ερώτησή μου είναι η εξής είναι απαραίτητο για να ικανοποιήσουμε, για να χαροποιήσουμε ε, τις, ε, τους οίκους αξιολόγησης να, ε, να έχουμε αυτήν την σχέση, αυτήν την αντίδραση σε σχέση με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών από τη στιγμή που στην αγορά υπάρχουν κάποια περίπλοκα τιμολόγια τα οποία αφορούν συγκεκριμένο τιμολόγιο το οποίο συνδέεται με κάποιο ειδικό πρόγραμμα πιστού καταναλωτή ας πούμε ε, και βάσει αυτού του συμβολέου δίνονται και κάποιες επιπλέον παροχές. Ερωτώ λοιπόν, οικονομικά ε, είναι χρήσιμο και ε, προσφέρει στην διαφάνεια να πρέπει να κάνουμε λογιστικές ακροβασίες οι οποίες τελικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και που στην ουσία κοστολογούν άμεσα ε, κάποια έσοδα τα οποία δεν θα μπορέσουν ουσιαστικά να ε, ληφθούν από τις εταιρείε τηλεπικοινωνιών παρά μόνο το τέλος της τιμολογιακής περίοδου και στο τέλος του συμβολέου. Νομίζω ότι μερικές φορές καλύτερα είναι να είμαστε πιο απλοί παρά να κάνουμε τα πράγματα πιο περίπλοκα. Απάντηση. Εάν ισχύει πραγματικά ότι ο καταναλωτής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, την επόμενη μέρα κιόλας που έχει υπογράψει το, συμβούλιο, το, ε, συμβόλαιο, να ακυρώσει το συμβόλαιο αυτό χωρίς καμία επιβάρυνση, τότε συμφωνώ απολύτως, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Εξάλλου είναι όλο και ε, είναι, ε, είναι σαφές ότι σε αυτή την περίπτωση καμία εταιρεία τηλεπικοινωνιών δεν θα έδινε αυτά τα δωρεάν ε, τηλέφωνα, αυτές δωρεάν τηλεφωνικές συσκευές, γιατί πλέον δεν θα ήταν οικονομικά αποδεκτό. Πάντως και το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο πολύ διαφορετικές τιμές, οι τιμολογήσεις είναι διαφορετικές. Ας πούμε να δέστε ένα iPad Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα λίγο πιο φτηνό, λίγο πιο, λίγο πιο ακριβό, αλλά στην ουσία ξέρουμε πόσο κοστίζει ένα iPad, όπως ξέρουμε και πόσο κοστίζει ε, ένα κινητό τηλέφωνο, μια συγκεκριμένη συσκευή. Το leasing, η χρονομίσθωση είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο λαμβάνουμε και εμείς υπόψη μας με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, εάν δει κανείς τα ε, παρελθόντα λογιστικά μεγάλα σκάνδαλα ε, στις ε, περισσότερες φορές αφορούσαν αυτά τα μυστικά κονδύλια και στην Ένρον στις Ηνωμένε Πολιτείε. Κάπου εκεί παίχτηκε το παιχνίδι γιατί ήταν εξαιρετικά προκλητικό για κάποιες εταιρείε να βάλουν πέραν των κανονικών λογιστικών λογαριασμών ορισμένες διαδικασίες στους ισολογισμούς τους δεν φαινόντουσαν αυτά τα περίεργα κονδύλια. Και πολύ συχνά αυτά τα συμβόλαια leasing είναι πάρα πολύ μεγάλα, μπορεί να αφορούν μακρές χρονικές περιόδους και επομένως θα πρέπει να φαίνονται σαφώς στον ισολογισμό. Είναι γεγονός ότι πολλές εταιρείες δεν συμφωνούν, δεν τους αρέσει και μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί πρέπει να, κατα... να αλλάξουν κάποιες διοικητικέ μεθόδους. Πάντως υπάρχουν και εταιρείε οι οποίες μας λένε ότι καταλαβαίνουμε τη θέση σας και συμφωνούμε γιατί οι επενδυτές θέλουν να βλέπουν αυτές τις πληροφορίες. Δεν θέλουν να αισθάνονται ότι ε, παρουσιάζουμε τα αριθμητικά στοιχεία με πιο αισιόδοξο τρόπο από ό,τι θα οφείλαμε. Μερικά σχόλια για ορισμένα από αυτά που είπατε σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και δεδομένου ότι με ακούσατε να σας αναφέρω για το τι κάναμε εκεί. Πρέπει να σας πω ότι ήμουν λίγο πιο απεσιόδοξη ε, σε ό,τι αφορά ε, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Γιατί έχουμε αλλάξει και λεξιλόγιο. Δεν λέμε ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε θα αλλάξουν τα πρότυπά του και θα έχουν το διεθνέ πρότυπο χρηματοοικονομική αγοράς. Αλλά μιλάμε για παράλληλη λειτουργία των δύο συστημάτων. Αυτό με ανησυχεί. Αλλά ελπίζω ε, ότι ήμουν επηρεασμένη από τη προηγούμενη γλώσσα που χρησιμοποιούσαμε. Σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα και κάποια άλλα, και για τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και για τις μεγαλύτερες, προβληματίζονται και το αφισβητούν, γιατί δεν μπορούν να ε, βλέπουν ε, πώς έχει η λειτουργία της επιχείρησης ε, Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ε, αυτό το παράδειγμα ε, για να κάνετε κάποιες προτάσεις έτσι για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αλλά αυτό είναι θέμα των εταιριών να το αποφασίσουν. Θα ήταν αυτό μια λύση. Απάντησε. Αυτό που χρησιμοποιούμε τώρα ως μέθοδος είναι πολύ κοινό ε, με το πρότυπο για το leasing. Δηλαδή, προσπαθούμε όσο γίνεται να αντικατοπτρίζουμε, να παρουσιάζουμε την οικονομική πραγματικότητα όπως έχει. Αλλά τη στιγμή που ο πελάτης παίρνει το κινητό τηλέφωνο, ε, αρχίζει να σκέφτεται ότι θα το αγοράσει και αρχίζει και καταβάλει ε, τις υποχρεώσεις του για επί ένα έτος ή δύο ε, με μορφή ενός τέλους. Αν δείτε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα Μπορεί κανείς να υπογράψει ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία χωρίς συσκευή ή με συσκευή κινητού τηλεφώνου και υπάρχουν και διαφορές ε, στις τιμές και στη τιμολόγηση και στο πώς ε, μετακυλούν ή συμπεριλαμβάνουν το κόστος του τηλεφώνου. Πάντως, ο καταναλωτής μπορεί την άλλη μέρα να επιστρέψει το συμβόλαιο να αρνηθεί και δεν νομίζω να υπάρχει πλέον ε, καμία διαφορά ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη. Για τις Ηνωμένε Πολιτείε γνωρίζω ότι διαφέρει το ύφο ανάλογα με ποιος είναι ο συνομιλητής σας. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα ληφθεί θετική απόφαση. Γιατί, διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επενδύσει πολλά τα πρότυπά μας στο Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και αν έπαιρναν ή αν πάρουν αρνητική απόφαση θα χάσουν την επιρροή τους στο δικό μας Συμβούλιο. Και δεν είναι προς το συμφέρον τους ουσιαστικά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ως επενδυτής ε, κάπου πρέπει να αποτανθεί. Ε, η Αμερική ανική αγορά δεν ανθεί και όλα σήμερα και όλοι γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη θα προέρθει από τις αναπτυσσόμενες, μάλλον τις αναδυόμενες αγορές. Ο Αμερικανός επενδυτής λοιπόν θα πρέπει να είναι σε θέση να ε, επαφίεται στη λογιστική αυτών των χωρών. Εξάλλου, γι' αυτό βγήκαν και αυτά τα πρότυπα μετά από το χάος στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην κρίση στην Ασία, όπου καταλάβαμε ότι ε, δεν ε, ήταν ε, συγκρίσιμα τα διάφορα λογιστικά πρότυπα που χρησιμοποιούσαν οι χώρες. Και επειδή εγώ πιστεύω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες ενδιαφέρονται να υπερασπιστούν τα οικονομικά του συμφέροντα, τελικά θα πάνε τη σωστή απόφαση. Thank you. Ευχαριστώ, Σβέν. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Έχω δύο σύντομα και ελπίζω συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα για το σχέδιο για τη δημιουργία των διεθνών προτύπων για την ε, για τις σηματοοικονομικές ε, εκθέσεις. Εκεί έχει αποσυρθεί το στοιχείο το οποίο αναφερόταν στην δημοσίευση των ε, επιτοκίων και των τόκων που πληρώνει κάποια επιχείρηση. Βέβαια, αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι δημόσια αγαθά τα λογιστικά αυτά στοιχεία θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για το ζήτημα αυτό, πόσο έχετε προχωρήσει στη διαδικασία διαβούλευσης για τα θέματα αυτά και ένα δεύτερο ερώτημα αναφέρεται σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα που είναι οι εκθέσεις κατά χώρα. Η πρόεδρος μας περιμένει να θέσω αυτό το ερώτημα εδώ και πολλή ώρα. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα θέματα αυτά το 2009 με τον προκάτοχό σας, τον κύριο Τουίντι, οποίος έκανε κάποια σχόλια για το θέμα αυτό, αλλά βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα και η Επιτροπή μας και η Ολομέλεια έχει πάρει μια θετική θέση για να υπάρχει μια παραγωγή εκθέσεων για κάθε χώρα μεμονωμένα. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξη, η κυρία Ζολή και εγώ ο ίδιος, είχαμε στείλει μια επιστολή στον προκάτοχό σας ζητώντας κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις για τα σχόλια που έκανε ενώπιον μας. Δυστυχώς ποτέ δεν πήραμε απάντηση. Αυτό με στενοχωρεί γιατί πιστεύουμε ότι <clears throat> εκεί υπάρχουν και κάποια προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ αρχών όπως η δική σας και εκλεγμένων κοινοβουλευτικών. Ο διάλογος σημαίνει ότι υπάρχει μια αμφίδρομη ροή πληροφορίας, θέτει κανεί ερωτήσεις, παίρνει απαντήσεις. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η δική σας θέση σε σχέση με την εφαρμογή στο IFRS, στο, στα πρότυπα χρηματοοικονομικών εκθέσεων, το να υπάρχει μια κατανομή αναχώρες και ελπίζω να μου δώσετε και μια έγγραφη απάντηση, ενδεχομένω με μορφή επιστολής. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ. Πρώτα απ' όλα, δεν νομίζω ότι αληθεύει ότι έχουμε χάσει τη δημόσια διάσταση της, του έργου μας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου εργαζόμενος για το δημόσιο συμφέρον. Πιστεύω ότι ακόμα εργάζομαι για το δημόσιο συμφέρον. Τι είναι το δημόσιο συμφέρον. Είναι ακριβώς το να υπάρξει μια προστασία του συμφέροντος των επενδυτών αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Φυσικά θα πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία τα οποία δίδουμε εμείς ως λογιστές για τις εταιρείε τις οποίες επενδύουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο επίπεδο δημοσίου συμφέροντος. Αλλά επειδή βρισκόμαστε και σε οικονομίες της αγοράς, δεν αρκούν μονάχα οι κανόνες, πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό λοιπόν το έργο μας για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις οικονομίες μας και στις αγορές. Και υπό την άποψη αυτή, η σωστή χρηματοοικονομική απεικόνηση μέσω εκθέσεων είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ε, σύγχρονης οικονομίας της αγοράς. Επομένως υπάρχει σημαντικό δημόσιο συμφέρον στο έργο μας <clears throat> και σίγουρα θα εξακολουθήσει να απεικονίζεται αυτό στα στρατηγικά μας έγγραφα. Εκθέσεις κατά χώρα. Έχω λιγότερη εμπειρία με το θέμα αυτό. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια τέτοια πρόταση θα χαρώ πολύ να δώσω μια απάντηση στην επιστολή σας και ξέρω ότι μόλις έχουμε δημοσιεύσει ένα έγγραφο διαβούλευσης για τη μελλοντική μας ημερησία διάταξη. Αναφέρεται το θέμα αυτό εκθέσεων κατά χώρα. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι θέλετε να κάνετε προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς έχουμε ήδη αποδειχθεί σε κάποια εργασία για τα θέματα αυτά η οποία δεν έχει υπερατωθεί. Ξέρω ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο <clears throat> και πολύ σημαντικό για το κοινοβούλιο σας. Υπάρχουν διάφοροι δρόμοι με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος σας, θα μπορούσε να γίνει με χρηματοοικονομικές εκθέσεις. Στις ΗΠΑ έχει περάσει αυτό μέσα από ένα αριθμιστικό πλαίσιο, αλλά μπορεί να επιτευχθεί ίσως και με άλλους τρόπους αυτός ο στόχος. Για μια ακόμα φορά όμως, η τελευταία μας στρατηγική ε, δήλωση λέει ότι πρέπει να υποστηρίξουμε το δημόσιο συμφέρον μέσα από τις ε, χρηματοοικονομικές λογιστικές απεικονίσεις. Αλλά με μεγάλη χαρά θα δώσω μια έγκαιρη απάντηση στην επιστολή σας. Ενδεχομένως ε, υπήρξε παρανόηση Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που αναφέρετε στη, στο έγγραφο στρατηγική σας και στις ε, αρχές ε, της αρχής της προτύπων. Εάν είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα ε, και αν θέλετε θα ήθελα να μου απαντήσετε. Ναι, είναι Ε, κοιτάξτε, εγώ είμαι κατά 99% σίγουρος ότι και στο αρχικό μας ε, πρόγραμμα γίνεται αναφορά στο δημόσιο συμφέρον. Ε, αν δεν γίνεται αναφορά, θα όφιλε να γίνεται. Pursued, I think the point is... Όπως ε, είπαμε και προηγουμένως στην κατηδία συνεδρία συζήτησή μας, ε, είναι ότι όσον αφορά αυτό το θέμα του, των λογαριασμών αναχώρα, ε, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου περάσει και η σχετική ρύθμιση και παρακαλούμε να το κάνετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Eh, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Δύο ερωτήσεις μόνο. Πρώτο, θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου ε, για την ε, συμπερίψη της ε, αναφοράς αναχώρα. Θέλουμε όλοι στο Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Χαίρομαι για τα διεθνή πρότυπα. Πριν από λίγα χρόνια μια μεγάλη γερμανική τράπεζα Όταν υπολόγιζε τα παράγωγά τη και την αξία του φαινόταν πενταπλάσια με βάση τα αμερικανικά πρότυπα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται και με το αρμπιτράζ ε, και ε, ποιε είναι οι αποκλήσει ε, στην μεταρρύθμιση αυτή τη χρηματοοικονομική και πώ θα τι υπερβούμε. Και ένα δεύτερο, αναφερθήκατε στα λογιστικά πρότυπα και την χρηματοοικονομική μεταρρύθμιση και κάτι άλλο που συνδέεται πάρα πολύ είναι η ε, ανάκαμψη της οικονομίας, γιατί ε, όλο αυτό συμβαδίζει με την ανάκαμψη οικονομίας και ε, Υπάρχουν και κάποιες ευαισθησίες. Τα νέα διεθνή πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν να έρθουν επενδύσεις και να τονωθεί η οικονομία, να σταματήσει αυτή η αστάθεια των αγορών. Αυτό μας ανησυχεί πολύ και, και να μην μεταφερθεί στα ενεργητικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Ε, γιατί αυτά είναι και μακροπρόθεσμα στοιχεία και μπορεί να προκληθεί κάποια στρέβλωση ε, των καταστάσεων εκεί. Και εσείς πώς θα προτίθεστε να τα ρυθμίσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Αναφέρατε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, στην καταγραφή, στα πρότυπα δηλαδή των Αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τα δικά μας. Είναι γεγονός αυτό. Και ποια είναι η βασική διαφορά. Στο διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αγοράς, όταν μια τράπεζα έχει μεγάλη παρουσία στην αγορά παραγωγών όπως οι περισσότερες, θα πρέπει όλα αυτά τα παράγωγα να τα έχουν στον ισολογισμό τους. Ε, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις ΗΠΑ οι θέσεις των παραγόγων ε, μπορούν να ισοσκελίζονται ενεργητικό και παθητικό. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ πιο περιορισμένο ισολογισμό. Και κατά μέσο όρο πιστεύω ότι αν οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπορούσαν να αντισταθμίζουν έτσι τα παράγωγα με τον τρόπο που το κάνουν στις ΗΠΑ οι τράπεζες, τότε οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπορεί να φαίνονταν 20 έως 30% μικρότερες ε, από ό,τι είναι σήμερα. Και για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι οι δικοί μας κανόνες είναι οι σωστοί. Διότι ένα στοιχείο ενεργητικού είναι συγκεκριμένο, ένα στοιχείο παθητικού είναι συγκεκριμένο. Και ε, τα παράγωγα είναι πολύ επικίνδυνα προϊόντα και δεν θα πρέπει να είναι κάπου στις υποσημειώσεις, αλλά στον ισολογισμό. Ε, πριν αναλάβω τη σημερινή μου θέση, ήμουν στην κεφαλαία αγορά της ε, Ολλανδίας. και ε, ένα μήνα πριν φτάσω, πάση περιπτώσει, ξέσπασε η χρηματοοικονομική κρίση. Δεν ε, λέω ότι συνδέονται αυτά, αλλά έψαχνα τι γίνεται στις οικονομίες μας, πού είναι τα ενεργητικά και είδα στατιστικές ευρωπαϊκών και αμερικανικών τραπεζών και φαινόταν σαν να υπήρχε πολύ μεγαλύτερη μόχλευση στην Ευρώπη από ό,τι στην Αμερική. Δεν ήταν αλήθεια αυτό. Όλοι είχαν πολύ υψηλή μόχλευση, αλλά επειδή τα αμερικανικά πρότυπα ε, είχαν αυτό τον τρόπο ε, υπολογισμού των παραγόγων ε, φαινόταν στα χαρτιά πολύ μεγάλη διαφορά. Και εγώ ήμουν ρυθμιστική αρχή. Υποτίθεται ότι παρακολουθούσα την αγορά με πολύ προσεκτικό μάτι. Καταλαβαίνετε το μέσο επενδυτή που δεν έχει όλες αυτές τις γνώσεις πόσο μπορεί να παραπλανηθεί και σοβαρά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα να συγκλίνει και είναι πολύ σημαντικό ακριβώ να έχουμε ένα είδος διεθνών προτύπων παγκοσμίω για να μπορεί ο κόσμος να συγκρίνει τη μία τράπεζα με την άλλη. Ε, Ανεξάρτητα από το που βρίσκονται. Το δεύτερο για την αστάθεια των αγορών. Όταν ήταν στο Ζενίθ η κρίση, ο μεγάλος πανικός, βέβαια θα μου πείτε και πότε ήταν στο Ζενίθ και τώρα που είναι, στο πρώτο εν πάση περιπτώσει, το 2008 μετά την κατάρρευση της τράπεζας ε, Lehman Brothers, πολλοί είπαν ότι η λογιστική ενίσχυε την κατάρρευση των αρκετών αγορών γιατί έδειχνε πόσο είχαν πέσει οι αξίες. Καταλαβαίνω ότι ε, επάνω εκεί στη βράση όλοι θεώρησαν ότι οι αγορές κατέρεαν. Αλλά εάν δούμε τώρα τι συνέβη και πώς είχαν οι λογιστικοί αριθμοί μετά το ξέσπασμα της κρίσης και τις πραγματικές απώλειες τελικά που υπομίστηκαν οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια, οι απώλειες αυτές ήταν πολύ μεγαλύτερες από ό,τι έδειχναν τα λογιστικά στοιχεία τότε στην αρχή της κρίσης. Λοιπόν, όχι απλώς δεν ε, το φουσκώσαμε, αλλά και ε, λίγα δείχναμε από αυτά που συνέβαιναν. Υπάρχει και ε, η έννοια στην οικονομία της αναμενόμενης απώλειας, αλλά αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν ότι ήταν μεγαλύτερες οι απώλειες από αυτές που φαινομενικά είχαν. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θα ήθελε να θέσει ερωτήματα. Ενδιαμέσως θα κάνω και εγώ κάποια ερωτήματα. Με ενδιαφέρε πολύ αυτή η συζήτηση που έγινε για την, ε, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η απεικόνιση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει χωριστούς, ε, χωριστές απεικονίσεις, χωριστές καταγραφές και γι' αυτό έχουμε το πλαίσιο αφαιρεγγιότητα 2 ότι είναι χωριστή λοιπόν η αντιμετώπιση των στοιχείων αυτών. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε κάποιο σημείο στο οποίο μπορεί να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού, όπως γίνεται στις ασφαλιστικές εταιρείες, όπου υπάρχει πράγματι κάποια σύνδεση μεταξύ κάποιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με κάποια έσοδα. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί για το θέμα αυτό. Και τώρα κάτι τελείως διαφορετικό, ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Στην ε, εισαγωγική σας ομιλία εσείς αναφερθήκατε ότι το γεγονός ότι, ότι δεν υπάρχουν πια στοιχεία ενεργητικού χωρίς καθόλου κίνδυνο, αυτό πάντα με ενδιέφερε σε ό,τι αφορούσε το κρατικό χρέος και τις απαιτήσεις, τις κεφαλουχικές απαιτήσεις για τις τράπεζες. Ίσως αυτό ήταν μία από τις αιτίε των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο κρατικού χρέους σήμερα. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε λιγάκι πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κανείς αυτό το πρόβλημα στα πλαίσια του δημοσίου χρέους των χωρών, ώστε να μην θεωρείται, ώστε να μην οδηγούμαστε σε μια υπερκυκλική αντιμετώπιση για, τα, για τις κεφαλουχικές απαιτήσει. Η αντιμετώπιση μέχρι στιγμής, όπως έχω δει, είναι είτε αλλάζει κανείς την στάθμιση κινδύνου, αυτό όμως μπορεί να είναι δύσκολο και να δημιουργεί προβλήματα. Ίσως μπορείτε να έχετε ένα ιδιαίτερο καθεστώς για τις μεγάλες εκθέσεις. Ξέρω ότι αυτό το θέμα δεν είναι αυτό το οποίο είναι η δικιά σας δουλειά, αλλά από λογιστική καθαρά πτυχή έχετε κάποιες ιδέες σε σχέση με το θέμα αυτό. Σίγουρα έχω ιδέες. Αλλά θα ξεπεράσω τώρα το, τα όρια μου ως αρμόδιος για τα λογιστικά πρότυπα. Αυτό που μου άνοιξε εμένα τα μάτια για το πόσο επικίνδυνα <clears throat> είναι τα συστήματα τα οποία θα ψηφίσετε σίγουρα σύντομα το CRD και το σύστημα στάθμισης κινδύνου της Βασιλείας είναι το παράδειγμα του τι έγινε στην Ιρλανδία. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια η Ιρλανδία δεν είχε καθόλου χρέος σε κρατικό επίπεδο, 23% μονάχα. Όλοι λέγανε ότι ήταν η πιο ασφαλής χώρα στην Ευρώπη και ήταν πραγματικά αλφα-αλφα-αλφα επίπεδου τα κρατικά αξιόγραφα. Είδαμε τι έγινε στη συνέχεια. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία ενεργητικού επενδυτικά ας πούμε, αξιόγραφα τα οποία να είναι απόλυτα ασφαλή. Θεωρείται τώρα η Γερμανία πιο ασφαλής, αλλά η Γερμανία έχει και αυτή 80% του ΑΕΠ χρέος, δημοσίου χρέος. Αν χρειάζεται να χρηματοδοτήσει <clears throat> μια μεγάλη ενέργεια διάσωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί το χρέος της να είναι πολύ πιο μεγάλο και στο μέλλον δεν θα μπορεί να παραμείνει σε επίπεδο 3α. Είδαμε τι έγινε και στι ΗΠΑ και αυτό ήταν αδιανόητο να υποβαθμιστεί η φεργιότητα των ΗΠΑ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο <clears throat> να έχουμε στον χρηματοπιστωτικό τομέα ένα καθεστώς το οποίο λέει για ότι ορισμένα είδη στοιχεία, στοιχείων ενεργητικού όπως είναι τα κρατικά αξιόγραφα ΑΑΑ δεν χρειάζεται να έχετε αποθέματα. Είναι μηδενική στάθμισή τους. Γι' αυτό πριν ξεκινήσει η τράπεζα, οι περισσότερε τράπεζε δείχνανε βάσει των κανόνων τη Βασιλεία να έχουν πολύ, υψηλά, πολύ ψηλό λόγο αποθεματικού κεφαλαίου. 10%, 11%. Αν χρησιμοποιούσατε όμω τα δικά μα λογιστικά στοιχεία, αυτά που δημοσιεύαμε εμεί, βλέπατε να έχουν ουσιαστικά 1% κεφάλαιο, κεφαλαιακό απόθεμα κτλ. Και αν αφορούσε κανείς τον, αναφερούσε κανείς τον αέρα και τους ε, μειοψηφούντες μετόχους, θα μπορούσαν να φτάσουν στο 0% ουσιαστικά. <clears throat> Αν θέλετε λοιπόν ένα απλό λόγο για το γιατί βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο μπάχαλο, είναι γιατί επιτρέψαμε στο χρηματοπιστωτικό τομέα να δουλεύει με μηδενικά περίπου κεφαλουχικά αποθέματα. Γι' αυτό το σύστημά μας είναι τόσο τροτό και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να έχουμε ένα σύστημα που μέσα στο οποίο επιτρέπεται να φερόμαστε σαν να μην υπάρχει κίνδυνο για ορισμένα στοιχεία ενεργητικού. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού έχουν κίνδυνο. Ναι, το άλλο ερώτημα τώρα. Αν υπάρχει στενή σχέση μεταξύ στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων παθητικού. Αν το λαμβάνει αυτό υπόψη βεβαίω. Ο κλάδο ασφάλεια ζωή, παραδείγματο τα προϊόντα ασφάλειας ζωής στην Ευρώπη, έχουν σαφή σύνδεση μεταξύ της, ε, του ασφαλιστικού συμβολέου που παίρνει κανείς ένα, μια απόδοση στην επένδυσή του αν η επένδυση την οποία έχει υποσχεθεί η εταιρεία σε αυτόν που έχει το ασφαλιστικό συμβόλαιο αν συνδέεται με την απόδοση των στοιχείων ενεργητικού στα οποία έχει επενδύσει η ασφαλιστική εταιρεία τα χρήματά της μπορεί να προκύψει ασφάλεια, γιατί όλα αυτά ανεβαίνουν και κατεβαίνουν μαζί. Ανεβαίνει η αγορά, ανεβαίνει η προσδοκόμενη απόδοση για τον ασφαλιζόμενο, πέφτει η αγορά, πέφτει και η απόδοση. Και ξέρουμε όταν θεσπίζουμε κανόνες λογιστικής, ότι αν υπάρχει μια στενή σύνδεση μεταξύ των στοιχείων παθητικού και των στοιχείων ενεργητικού, δεν πρέπει να υπάρχει έλλειψη αντιστοιχία σε λογιστικού όρου. Ευχαριστώ πολύ. Καμιά άλλη ερώτηση, κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Όχι, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Δεν ξέρω, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αν θέλετε κάτι να πείτε ή εσείς αν θέλετε να ολοκληρώσετε. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει λείψει τίποτα. Ε, νομίζω ότι έχουμε κάνει το γύρο του κόσμου και έχουμε αναφερθεί στα πιο σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα πάντως ε, να σας ευχαριστήσω για την προσοχή που δείξατε. Με μεγάλη μου χαρά θα επανέλθω έτσι ώστε να συζητήσω μαζί σας και βεβαίως ε, ό,τι ερωτήματα έχετε μπορώ να τα πάρω μαζί μου και να απαντήσω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ. Um, we've got about a, ε, λοιπόν, θα κάνουμε δεκάλεπτη, ένα δεκάλεπτο διάλειμμα πριν από την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ πολύ.

Okay, everybody. Ωραία λοιπόν, νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Ε, δεν έχει έρθει ακόμα ο Γκέι Μίτσελ. Αργοπόρησε λίγο, δεν ξέρω. Oh, are you speaking on behalf of... you have a coordinator. Well... Έχουμε εδώ λαμπρό συντονιστή, δεν έχουμε πρόβλημα. Right, oh, and I'm, I'm, I'm Okay. Um, and we are also missing... Μας λείπουν και άλλοι όμως. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι θα έρθουν ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η εξέταση των ε, τροπολογιών. Θα δώσω τον λόγο στο Ραμόν, τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι γιατί οι περισσότεροι μεταξύ ημών ε, ε, μελετήσατε προσεκτικά την έκθεση και έχουν υποβληθεί πάρα πολλές τροπολογίες. Ε, πιστεύω ότι με συνεννόηση και καλή θέληση υπάρχει τρόπος και χώρος για ε, συμβιβασμούς. Η συζήτηση ήταν πλούσια. Ξέρετε ότι αυτή η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ε, σημαντική. Ε, ποιοι από εμά και πόσοι ε, μπορούσαν να φανταστούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ήταν υποχρεωμένη να αγοράσει ομόλογα. Ε, ξεπέρασαν και τους χειρότερους εφιάλτες μας τα πράγματα και η κατάσταση και επομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπρεπε να δείξει πολύ καλό τιμόνι. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ε, χωρίς την παρέμβαση που έγινε ας πούμε, τον προηγούμενο Αύγουστο στις αγορές η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη θα πρέπει να υπάρξει νέο πλαίσιο που θα ελαφρύνει το βάρος αυτό από, τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα πρέπει ε, να ε, υπάρξουν αυτά τα θεσμικά όργανα τα οποία θα δημιουργήσουν τους νέους οικονομικούς οργανισμούς που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να βγει όσο γίνεται πιο γρήγορα από την ε, οικονομική κρίση. Όσον αφορά την απόδοση και την επίδοση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, ε, συμφωνούμε με τους ε, ΕΛΚ, σοσιαλιστές και πρασίνους, ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι προσωρινά, έστω και αν ήταν απαραίτητα αυτή την περίοδο της κρίσης. Συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να παραμείνει πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά τα παράπλευρα ε, και ότι και και τις εγγυήσεις ε, και ε, ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Ο κύριος Γκάι Μίτσελ, ο σκιώδης ηγητής, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι εδώ, με βρίσκει σύμφωνο με τις απόψεις που έχει εκφράσει. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ασκήσει δημοσιονομική πολιτική και να εισπράξει φόρους με τους σοσιαλιστές και τους δημοκράτες, κυρίως δεν με τον κύριο Κούτας, συμφωνούμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει ε, στον δρόμο της ολοκλήρωσης. Ε, είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να ότι δεν, δεν εννοούμε τα ίδια πράγματα όταν μιλάμε για εγγύησεις και για ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Ε, οι πράσινοι επίσης έχουν ε, πάρα πολύ σωστές απόψεις και συμφωνώ μαζί τους όσον αφορά την τεχνογνωσία και την διαφάνεια. Ε, Σβέν, θα, συμφω... θα εγγράψω πολλές από τις τροπολογίες σου γιατί με βρίσκουν σύμφωνο και χαίρομαι που έχουμε την ίδια άποψη όσον αφορά την μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τον στόχο 2. Τέλος, όσον αφορά τι τροπολογίε της ΓΟΕ, πρέπει να πω ότι έστω και αν έχουμε πολύ διαφορετική ιδεολογική αρχή σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε σε θέματα επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ας πούμε, τον ε, ρόλο της χρηματοοικονομικής πολιτικής στην δημιουργία ε, νέων ε, όσον αφορά τις φούσκες τις οικονομικές, ε, το θέμα της ε, διαφάνειας Τώρα ε, υπάρχουν ε, κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες με βρίσκουν σύμφωνο, λέω τροπολογίες οι οποίες δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν ορισμένα πρακτικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως άλλωστε γίνεται και σε πάρα πολλές άλλες χώρες μεταξύ των οποίων στην Ιαπωνία και στην Ελβετία. Πολλές φορές διαβάζω ότι ε, διαβάζω ότι σε πολλές περιπτώσεις ε, δεν πρέπει τα πρακτικά να δημοσιοποιούνται, αλλά πιστεύω ότι σε μερικές περιπτώσεις, όπως ας πούμε τον προηγούμενο Αύγουστο που είδαμε ότι ε, κάποιοι από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν συμφώνησαν με, την, με τα σχέδια διάσωσης της Ιταλίας ή άλλων χωρών. Διαβάσαμε όμως τελικά γιατί διέρευσαν στον τύπο ε, κάποια από τα στοιχεία της συζήτησης. Ίσως δεν ήταν καλύτερο ε, να ε, υπάρχει δημοσίευση των πρακτικών έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς και ποια ήταν η επιχειρηματολογία η οποία ε, οδήγησε εις ε, τη λήψη των αποφάσεων. Επίσης, η δημοσιοποίηση των πρακτικών ε, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τους οικονομικούς παρατηρητές για πληρέστερες οικονομικές προβλέψεις. Επίσης, οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μην ξεχνάμε ότι παραμένει το κεντρικό οικοδόμημα, ο κεντρικό θεσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα οικονομικά. Ε, είπα και προηγουμένω ότι θα έρθω σε επαφή με του σκιώδε συγητέ, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε κάποιε συμβαστικέ ε, ε, λύσει και βεβαίω ε, οποιοδήποτε θέλει περαιτέρω πληροφορία όσον αφορά την έκθεση αυτή μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μου. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σα για περαιτέρω συζητήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούτες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω επαναλαμβάνω για και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τρέμολς, ότι το ο κύριος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή επίλυση της κρίσης που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια κρίση η οποία πρέπει να εξασφαλίσει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό έχω καταθέσει μια σειρά από τροπολογίε για να μπορέσουμε να δείξουμε μια θετικότερη ενατένση για τον χώρο τη Ευρωζώνη και να έχουμε ένα πιο στεναρό μήνυμα για μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Εγώ χαιρετίζω την ε, παρουσία τη ΕΚΤ για την αντιμετώπιση τη ε, χρηματοπιστωτικής κλίσης και τη κρίση κρατικού χρέου, αλλά χρειάζεται και μια πιο μακροχρόνια λύση. Αυτό απαιτεί και μια ένωση σε επίπεδο φορολογικό, έκδοση ευρωομολόγων κτλ. Για τις τροπολογίες που έχω καταθέσει εξ ονόματος της ομάδας μου, θα ήθελα να πω ότι αυτό το που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε την ευρωστία της ζώνης του ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια σειρά ε, μέτρων και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο ε, εργασιακής αγοράς ώστε να υπάρξει μια μεγαλύτερη δυνατότητα συντονισμού, να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρξει λοιπόν ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός ο οποίος θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά και πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο προς την κατεύθυνση συμβαστικών λύσεων και είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν καταθέσει τροπολογίες. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ήδη αυτή τη βδομάδα τις συμβαστικές τροπολογίες του εισηγητή, είπε αύριο ή μεθαύριο και μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια καλή συζήτηση μαζί του μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρώτα, πρώτα οι σκιώδεις συζητητές, Σίλβι, αν θες. Ο Σβέν πρώτα. Ευχαριστώ, Ραμόν, για την έκθεσή σου και τις διευκρινήσεις που μας έδωσες. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή συμφωνία μεταξύ των τροπολογιών. Υπάρχουν κοινέ κατευθύνσεις σε πολλές από αυτές τις τροπολογίες. Έχουμε τώρα πολλά από τα συνηθισμένα θέματα, τα οποία πρέπει να καλύψουν οι συζητήσει μα για τις συμβαστικέ τροπολογίες. Ένα από αυτά τα θέματα που είναι σημαντικό για μένα, το ανέφερε στην αρχή, είναι η σημασία τη νομισματικής πολιτική για τη δημιουργία φυσαλίδων που να βασίζονται σε στοιχεία ενεργητικού. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να συζητήσουμε πολύ περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξέρουμε ότι δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό της ε, σταθερότητας των τιμών, που είναι ο κύριος στόχος της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά τα μακροχρόνια αποτελέσματα των ε, χαμηλού επιτοχίου δανείων οδήγησαν στη δημιουργία φουσκών που βασίζονται παραγωγικά στην κατασκευαστική ε, αγορά, στην αγορά που βασίζεται σε στοιχεία ενεργητικού. Επομένως θα πρέπει και εδώ να βρούμε μια σαφή διατύπωση. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες, όπως και αυτή του κ. Σιούτας, οι οποίες ζητούν να λάβουμε υπόψη και τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Που είναι μια άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Υποστηρίζω επίσης αυτά που είπες για τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και πιστεύω ότι η τροπολογία της Σιλβί Γκουλάρ πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν αφορά μόνο τα πρακτικά Πρόκειται για την ε, ποιότητα των εγγυητικών στοιχείων. Είχαμε αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Τρισέ. Είπε ότι μόνο ένα τμήμα του, του ενέχειρου των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για εγγύηση χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας. Βέβαια, το θέμα του συνολικού ποσού για την εγκυοδοσία δεν έχει μεγάλη σημασία για την ε, φερεγγιότητα μεμονωμένων πιστοτικών ιδρυμάτων. Προφανώς προκύπτουν λοιπόν ερωτήματα και από τη δική μας άποψη τα πράγματα δεν είναι τόσο διάφανα όσο θα πρέπει να είναι για το τι γίνεται αποδεκτό ως ε, εγκυοδοσία <clears throat> από την Κεντρική Τράπεζα και πώς γίνονται απομειώσεις σε σχέση με την ονομαστική αξία των εγκυητικών αυτών των εγγύησεων αυτών. Και εδώ έχουμε μια σειρά από ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ευαισθησία που επιδεικνύει σε σχέση με σφάλματα στην αξιολόγηση, στην εκτίμηση των αξιών των εγγύησεων. Θα σταματήσω εδώ, αλλά έχω ακόμα ένα σημείο το οποίο θέλω να θίξω, το οποίο και αυτό είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας. Και εδώ το συμμεριζόμαι απόλυτα με τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγκάστηκε να αναλάβει πολλές λειτουργίες που δεν προβλεπόταν να τις επομιστεί και υπάρχει μια μεγάλη τάση σε πολλά κράτη-μέλη να πούν δεν μας αρέσει να πάρει αυτές τις αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά δεν θέλουμε και οι κυβερνήσεις να συνεργαστούν και να βρουν αυτές οι κυβερνήσεις μια λύση για τα θέματα αυτά. Δεν πρέπει να πέσουμε λοιπόν σε αυτή την παγίδα. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τις κύριες λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια. Χρειαζόμαστε μια βαθύτερη φορολογική <clears throat> και δημοσιονομική ένωση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εσύ αναφέρει τα κύρια συστατικά μια τέτοια ένωση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επομένω αυτή την έκθεση για να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Αλλιώ αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια ατυχή θέση όπου έχει υποχρεωθεί να παίρνει αποφάσεις που δεν προβλεπόταν να τις παίρνει αυτή και για τις οποίες απαιτείται και μια μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Για μένα αυτό είναι το κύριο λοιπόν θέμα που έχει να κάνει με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς το παρόν και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή δήλωση από τη δική μας πλευρά. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τα προβλήματα, αλλά η απάντηση στα προβλήματα αυτά δεν είναι να ρίξουμε το φταίξιμο στην ΕΚΤ. <clears throat> Αντίθετα, θα πρέπει να ανακουφίσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το να πάρουν τις αρμοδιότητες αυτές οι κατάλληλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι πρόκειται για την ετήσια έκθεση για το 2010 ε, η έκθεση δική μας για την έκθεση της ΕΚΤ, εν περιπτώσει, το έχουμε διευρύνει ε, ε, ε, θα πρέπει να είμαστε πολιτικοί ε, στη σκέψη μα αυτή τη στιγμή, λέει ο κύριο Γκίγκολτ. Ναι, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον, ε, λέει ο πρόεδρο, αλλά την άλλη φορά να αλλάξουμε τον τίτλο. Να μιλάμε και για ανταγωνισμό. Κύριο Χουντή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή, ε, καθώς από την προφορική του σημερινή παρουσίαση έδειξε ένα πνεύμα συνεργασίας αυτό θα το αξιοποιήσουμε και εμείς προσπαθώντας να αξιοποιηθούν οι δικές μας οι τροπολογίες. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι, επειδή αναφέρθηκε για άλλη μια φορά ο εισηγητής σήμερα, ότι οι τροπολογίες μας δεν ξεπηδάνε, δεν προκύπτουν από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές που έχουμε γενικώ ή και ειδικά για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τουλάχιστον αρκετές από αυτές. Βγαίνουν από την εμπειρία και από αυτό που θέλουμε να εκτιμήσουμε με τη δική μας έκθεση σχετικά με τα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το προηγούμενο έτος, που είναι και το αντικείμενο της έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προηγούμενο έτος και σήμερα που έχουμε μπει στο 2011 στα γεμάτα, είμαστε σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη μια διευρυμένη κρίση όπως και να το πει κανείς, της Ευρωζώνης. Είναι άδικο, συμφωνώ, να βάλουμε όλα τα προβλήματα ως ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι άδικο. Και βεβαίως δεν μπορεί να τις βάλει σε όλα τα, τα προβλήματα. Αλλά με τις τροπολογίες, δύο-τρία θα πω εγώ ακόμα, υπάρχει ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε αρκετές χώρες και συνολικά στην Ευρωζώνη. Και αυτό έχει επισημανθεί από τις παρατηρήσεις της ε, δικές μας. Η βασική παρατήρηση είναι ότι όσο εκ του καταστατικού, εκ της δομής της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός δανεισμού τελευταίας καταφυγής σε περιπτώσεις γενικότερης ή τοπικής κρίσης, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ουσιαστικά. Ορισμένα τα προβλήματα ήδη επισημαίνονται και από τον εισηγητή και από άλλους συναδέλφους με την έννοια της προτροπής για να ληφθούν κάποια μέτρα και με τα οποία, τα οποία στηρίζουμε και τα οποία θα υποστηρίξουμε σε σχέση με τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει άλλοι συνάδελφοι. Αναφέρομαι σε δύο. Σχετικά με το τι θα γίνει επιτέλους με τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης εδώ το κακό είναι ενώ αποδοκιμάζονται, ενώ καταγγέλλονται, δεν λαμβάνονται μέτρα να περιοριστεί αυτή η καταστροφική δράση της. Ο εισηγητής το αντιλαμβάνεται, γι' αυτό προτείνει κάτι διαφορετικό. Το έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές. Αλλά αυτή η ανοχή βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, κάθε φορά με τις παρεμβάσεις, με τις υποβαθμίσεις και ούτω καθεξής. Δεύτερον, βεβαίως υποστηρίζουμε την ιδέα για το ευρωομόλογο. Κουβεντιάσαμε και ως προς αυτό. Αλλά ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι, ορισμένα και σωστά μέτρα όταν καθυστερούν να παρθούν, καθυστερούν να λυθούν, είναι ανεπαρκή στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος που έχουμε ως προς ε, το, το θέμα αυτό που κουβεντιάζουμε. Βεβαίως, εντάξει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει ο καταστατικός στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή να έχει σαν μόνο, μόνο, στόχο τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει εποφελία. Αλλά αυτό το αντιλαμβάνομαι ότι θέλει μεγάλη συζήτηση, δεν απαιτώ ότι πρέπει να είναι <laughs> από αυτά που θα συμφωνήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ορισμένε από τι ενστάσει μα προσπάθησα να τι αναφέρω σύντομα. Ε, ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη διάθεση για συνεργασία και θα επιχειρήσουμε στι συμβιβαστικέ προτάσει να μπουν και ορισμένε από τι δικέ μα ιδέε για να δούμε ένα καλύτερο, όπω πιστεύουμε, αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σίλβε Γκουλάρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σύντομα, δύο μόνο πράγματα, γιατί ο εισηγητή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά αφενό και πετέρου έχουν υποθεί πολλά ήδη. Θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό που είπε ο Σφέν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να ε, ειδωθεί αποκομμένη ε, στο γενικό σύνολο στην κοινότητα και αυτό είναι ο κίνδυνος σε αυτές τις εκθέσεις. Σήμερα αναγκάστηκε να κάνει κάποια πράγματα που δεν είχαν προβλεφθεί πάρα πολύ. Εδώ στις 29 Αυγούστου μας το είπε και ο κύριος Τρισέ λόγω της αδράνειας κάποιων άλλων θεσμικών οργάνων. Είναι σημαντικό λοιπόν να το τονίσουμε αυτό. Μας ενδιαφέρει να βρούμε μια σωστή λύση ε, προς όφελος της Ευρώπης που να διαφυλάσει την αποστολή της ΕΚΤ χωρίς να, αφήνει, να δημιουργηθεί κενό. Μια μικρή ερώτηση για τα θέματα της διαφάνειας και το έχω συζητήσει με τον Γαμόν. Όταν ε, συγκρίνουμε τα όσα ε, συμβαίνουν στην Ευρωζώνη με άλλες κεντρικές τράπεζες, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα το εξή στοιχείο. Και στη ΣΥΠΑ και στην Ιαπωνία και αλλού είναι ένα το νόμισμα και ένα το χρέος. Και όταν κάποιος κυβερνήτης ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής του Τράπεζας από την Καλιφόρνια, από την Εμπράσκα, και ε, βγει και πει κάτι και δηλώσει, αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τα spreads στις ΗΠΑ. Εγώ βεβαίως είμαι ε, υπέρ Τη διαφάνεια και πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε απόκληση θα μπορούσε ε, να ε, είναι μπαλάκι στα χέρια των αγορών ε, που να φέρνουν τη μία χώρα απέναντι σε μια άλλη και τα λοιπά με κάποιες προβολές και με κάποιες προεκτάσεις. Αυτό λίγο με ενοχλεί, γιατί θα είναι παράγον διχόνοιας που θα στραφεί κατά της Ευρωπαϊκής Συνοχής και θα έχει και συνέπειε που δεν υπάρχουν εκ των πραγμάτων και εκ της πίσω με άλλα συστήματα με τα οποία συγκρινόμαστε. Mm. Άλλος κανείς. Ο Αλλά όχι, Άστριτ προηγουμένω, συγγνώμη. Ναι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Λούλινγκ. Πρέπει να σας πω ότι δεν είχα ακόμα ασχοληθεί με την έκθεση αυτή, γιατί είχα άλλε προτεραιότητε αυτόν τον καιρό, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις Μόλις διάβασα στον τύπο, αλλά δεν το βρίσκω που το διάβασα, ότι κάποιος Γερμανός θέλει να προσφύγει κατά του κυρίου Τρισέ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω υπέρβασης καθηκόντων. Αν δεν απατώμε αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ερωτήσεις στον κύριο Τρισέ ε, ε, για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό το διάβημα του Γερμανού, πώς να το χαρακτηρίσω. Αυτά δεν μας καθησυχάζουν. έκαθεν εγώ υπερασπίστηκα τον κύριο Τρισέ και έλεγα ότι ήταν ο μόνος που δρούσε όταν όλοι οι άλλοι ήταν απόντες. Έλαμπαν δια της απουσίας τους, σε πάση περιπτώσει, οι Κομισιόν και άλλοι, όταν οι κυβερνήσεις και κάποιες πρωτεύουσες είχαν, πώς να το πω για να παραμείνω ευγενική, ε, ε, ανέλαβαν κάποιες πρωτοβουλίες ε, που καλά θα ήταν να μην είχαν αναλάβει. Ο σκιώτης ηγητής μας έχει τροπολογίες. Αν ήταν εδώ ο κύριος Γκαρσία Μαργκάγιο θα έχει πάρει και το λόγο σίγουρα. Αλλά θέλω να ρωτήσω. Τι θα κάνουμε. Καλεί ο εισηγητής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει ένα ευρωπαϊκό οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ε, ο κύριος Μίτσελ θέλει να το καταργήσει αυτό. Μόλις διάβασα δε στο γερμανικό τύπο ότι τώρα έρχεται ο κύριος Γκίντο Βέστερβέλε, υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας και γράφει άρθρα στον τύπο και ζητάει και αυτός ένα οίκο αξιολόγηση. Θέλω να ρωτήσω τον εισηγητή τι πιστεύει. Πραγματικά αυτό μας χρειάζεται τώρα, ένας ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Σπεν, got a little comeback on something. θες να επανέλθεις λίγο σε κάτι. Πάρα πολύ σύντομα. Αγαπητή κυρία Λούλινγκ, μην τα παίρνετε σοβαρά όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία. Αυτό ισχύει και για τις μόνιμες προσφυγές σε διάφορα δικαστήρια κατά ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή ε, ε, ευρωπαϊκών συνθήκων το θέμα του Ευρωπαϊκού Οίκου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι στο συμβόλαιο, στη συμφωνία του συνασπισμού που κυβερνάει στη Γερμανία, αλλά μέχρι τώρα ποτέ δεν το έχουν συγκεκριμενοποιήσει. Ποιο μοντέλο θα έχει, πώς θα λειτουργεί, εδώ και καιρό το περιμένουμε αυτό. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση του Wolf Klintz ζητήσαμε ένα ίδρυμα τέτοιο να ε, δημιουργηθεί ε, Τότε αυτό διαγράφει. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτό, ούτε με ικανοποίησε. Τώρα έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα. Και ακούω, με, με έκπληξη, επαναλαμβάνω, με έκπληξη ακούω, ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ ασαφές το πράγμα. Για τον επόμενο γύρο μεταρρυθμίσεων στους οίκους αξιολόγησης, εάν θα συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους και αυτή θεωρώ ότι είναι σωστό να το αναφέρουμε και να πούμε ότι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κοινή θέση. Όχι γιατί λέμε ότι όλα θα πρέπει να είναι στα χέρια του δημοσίου, αλλά εκτός από τη χρηματοδότηση, εκείνοι που εκδίδουν ε, αξιόγραφα ε, είναι μια ιστορία, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι φορεί για να είναι μεγαλύτερη ποικιλία στι αγορέ. Γι' αυτό ζητάμε ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα αξιολόγηση και θεωρούσα ότι εδώ και καιρό είχαμε αυτή τη θέση. Αν τώρα ο κύριος Βέστερ θα μπορούσε να συμβάλλει η κυβέρνηση επιτέλους να κάνει και δική της πρόταση, τότε θα τον ε, λάμβανα πιο σοβαρά υπόψη τουλάχιστον σε αυτό. Okay, I Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει τους ομιλητές. Μόνο ο Ραμόν έχει να απαντήσει μονάχα και του ξαναδίνει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Για τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης. Μια ενδεχόμενη λύση θα ήταν να εισαγάγουμε και μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Δεν είμαι εναντίον των φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, έχουν ένα ρόλο διαδραματίσουν που είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ τους και θα πρέπει να είναι λιγότερο πολυδάπανες οι υπηρεσίε τους επίσης. Ένας τρόπος να το επιτύχουμε αυτό είναι να δημιουργήσουμε και ένα δημόσιο φορέα πιστοληπτικής αξιολόγηση, ο οποίο και αυτός θα μπορούσε να παίζει ένα ρόλο σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι ο κύριος Κλίντς <clears throat> έχει δίκιο. Γιατί να μην ακολουθήσουμε την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια οι φορείς αυτοί, οι δημόσιοι, δεν θα μπορούσαν να είναι οι πιο πρόσφοροι για να πούν αν το δημόσιο χρέος μιας χώρας είναι πιο βαρύ από το χρέος μιας άλλης χώρας, αλλά αυτό θα ήταν ένας τρόπος να εισαγάγουμε περισσότερο αναγωνισμό στον τομέα αυτό και θα ήταν θετικό και για τις αγορές. και όπως είπα στην παρουσίαση της έκθεσης, εγώ συνέγραψα αυτή την έκθεση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μέσα στο... στην κρίση που αντιμετωπίσαμε το καλοκαίρι και έχω γράψει αυτή την έκθεση ως μεσογειακός αλλά και φιλελεύθερος. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση γιατί δεν είμαστε πολύ μεσογειακοί φιλελεύθεροι σε αυτή, την αίθουσα και σε αυτό το κοινοβούλιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όμως να σταθούμε στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και για τα οποία μας ζητούν να δώσουμε μια λύση. Νομίζω ότι είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παίζει πια ένα ιονί δημοσιονομικό ρόλο. Και φυσικά δεν ήταν προετοιμασμένη να κάνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να βελτιώσουμε το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να απαλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την ανάγκη να παίξει αυτό το ρόλο. Αν δεν απατώμε, νομίζω ότι ο Επίτροπος ολιρέν, το Μάιο του 2010 είχε προτείνει <clears throat> να δώσουμε εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να αγοράζει ομόλογα στη δευτερογενή αγορά για να διατηρήσει τις τιμές τους σε σωστό επίπεδο. Εμείς είπαμε όχι τότε όμως. Και επειδή δεν υπήρξε μια τέτοια ευρωπαϊκή λύση, είμαστε επί ξηρού ακμής. Όλο αυτό το καλοκαίρι βρεθήκαμε επί ξηρού ακμής και δεν ξέρουμε τι μέρα θα ξημερώσει στις αγορές αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρξει ε, πάυση πληρωμών σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή αποτελεί και μια ευκαιρία να συζητήσουμε για την ε, Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Ένωση που χρειαζόμαστε για το ελάχιστο επίπεδο ολοκλήρωση στο δημοσιονομικό τομέα που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει. Πιστεύω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι ότι πρέπει να έχουμε μια πραγματιστική προσέγγιση στα θέματα αυτά, κάτι το οποίο θα διευκολύνει και την επίτευξη κοινών θέσεων, θέσεων κοινή υποστήριξη, κάτι που θα δώσει ένα σαφέ μήνυμα και προ το Συμβούλιο και προ την Κομισιόν και στον Ευρωπαίο πολίτη ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους να λύσουμε αυτή την κρίση και να αποτρέψουμε και τις επόμενες κρίσεις. Για τη Σιλβή τώρα, για τα πρακτικά. Έχεις δίκιο Σιλβή. Μπορεί να είναι ένας παράγων διχόνοιας Και εγώ αναρωτιέμαι. Η μη δημοσίευση πρακτικών είναι μήνυμα αδυναμίας σε επίπεδο της ε, ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μια νομισματική ένωση η οποία για μένα ως φιλελεύθερο από τη Μεσόγειο ήταν ένα ασφαλές αγκυροβόλιο. Ήταν αυτοίστημα χωρίς το οποίο η Ισπανία θα είχε υποφέρει πολύ περισσότερο. Κάθε μέρα που ξεκινάω τη μέρα μου λέω ευχαριστώ νομισματική ένωση. Ναι, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, αλλά ως φιλελεύθερος από τη Μεσόγειο το ξαναλέω κάθε μέρα. Καλά που υπάρχει η νομισματική ένωση. Αυτή την ένωση λοιπόν που έχουμε δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Αλλά μια τέτοια ένωση δεν θα πρέπει να έχει αντιρρήσει για τη δημοσίευση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό εγώ επανέλαβα αυτά τα επιχειρήματα για τη διαφάνεια. ούτω, ή άλλω θα τα συζητήσουμε, θα τα ψηφίσουμε και θα βγει από εμά ένα μήνυμα σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε στις 11 Οκτωβρίου και ο στόχος μας είναι να φέρουμε το θέμα στην Ολομέλεια στις 2 Νοεμβρίου στη δεύτερη μάλλον ολομέλεια του Νοεμβρίου. Κλείσαμε λοιπόν τη συζήτηση για την ε, ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τίποτα άλλο δεν έχει ημερησία διάταξη. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν νωρί την συνεδρίασή μας, εκτός αν κάποιος θέλει να θίξει κάποιο ζήτημα. Αυτή είναι η ευκαιρία σας. Όχι. Ωραία. Μπορούμε να κλείσουμε νωρί και όχι αργά. Πολύ ωραία. Αν δεν πειράζει που ήρθες τώρα, δεν το κάνουμε επίτηδες.